για την κατάσταση στις Μαλτίβες. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Μίμητ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, κύριε και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση των Μαλτιβών έχει αναλάβει σημαντικά βήματα για νομοθεσία κατά της οικίας βίας, τη διακίνηση ανθρώπων, το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την βελτιωμένη κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει τα μέτρα αυτά. Όμως αυτά τα βήματα μπορεί να υπονομευθούν εφόσον η κυβέρνηση δεν αναλάβει κατεπίγουσα δράση για να αποκαταστήσει την υγεία του δημοκρατικού καθεστώτος και την ε, προστασία βασικών ε, δημοκρατικών αξιών από των οποίων θεμελιώνεται το δημοκρατικό σύστημα. Οι Μαλδίβες είναι μια νέα και ευάλωτη δημοκρατία από την έγκριση του νέου συστήματος, συντάγματος και τις πολυκομματικές εκλογές το 2008 έχει επιτευχθεί πρόοδος αλλά άνηση. Ιδίως ε, μετά την ε, αμφιλεγόμενη αλλαγή εξουσίας το Φεβρουάριο 2012 οι διακλαδώσεις ε, και οι επιπτώσεις αυτών των γεγονότων υπονομεύουν τις πιθανότητες προόδου και εκδημοκρατισμού των Μαλτιβών. Ο πρώην πρόεδρος Νασίντ στις 22 Φεβρουαρίου φέτος ε, οδήγησε και ενέτεινε Ε, προκάλεσε προκάλεσε επεισόδια και συνελήφθη. Ε, στην ε, Ελβετία εκφράστηκαν ανησυχίες για τη σύλληψη και την ε, συμπεριφορά αυτή στην πρώτη ε, εκδίκαση που έλαβε χώρα χωρίς καμία παρουσία συνηγόρου. Μετά την καταδίκη σε 13 χρόνια κάθυρξη στις 13 Μαρτίου φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έκανε δήλωση με σοβαρά ερωτήματα για την σοβαρές απορίες για την, ε, υπονόμευση, για την κατάσταση του δικαστικού συστήματος και το κατά πόσο μπορούν οι πολίτες να το εμπιστεύονται. Οι δηλώσεις αυτές τονίζουν την ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών αρχών για το Σύνταγμα, για το κάτος δικαίου, για τις ε, ένομες διαδικασίες και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Θέλω λοιπόν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τονίσω και επαναλάβω την σημασία των αρχών αυτών. Οι αρχές αυτές είναι θεμελιώδεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι για να ε, προστατεύσουμε τις ένομες ε, ελπίδες των ανθρώπων αυτών για εκδημοκρατισμό στις Μαλδίβες ε, και ανά τον κόσμο. Οι ε, πολίτες των Μαλδιβών δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους. Πρέπει να λάβουμε δράση τώρα για να δείξουμε την αφοσίωσή μας στην ελευθερία της έκφρασης και του συγκεντρώνεστε. Η αρχές, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους ε, χωρίς ε, να καταπιέζονται από τις αρχές του κράτους και στις Μαλδίβες και ανεξάρτητα σώματα όπως η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι εκλογικές, οι Επιτροπέ επιτροπές έχουν ε, καθοριστικό ρόλο διαρματίσουν στη διατήρηση του δημοκρατικού καθεστώτος. Επιτρέπουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα και αρμοδιότητες να, ε, να έρχονται εις πέρας χωρίς να φοβούνται ότι θα επιβληθούν κυρώσεις ή ποινές. Και επίσης θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται δημοκρατικά και η δράση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να επιβάλλει νομικούς περιορισμούς περιορισμού στην ελευθεροτυπία ή την ελευθερία έκφραση των μέσων μαζική ενημέρωση. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οποιαδήποτε ε, καταστολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, ε, ερευνάται και έρχεται ενώπιον της δικαιοσύνης. Είπατε εκπρόσωπο και αντιπρόοδος έχει λάβει έτοιμα από την κυβέρνηση των Μαλτιβών να αποσταλούν παρατηρητές για την εξέταση της αίτησης του κυρίου Νασίτ. Η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόοδος έχει προσφερθεί να στείλει νομικό εμπειρογνώμονα όχι μόνο για να εξετάσει την υπόθεση Νασίτ αλλά και για να βοηθήσει στην αναθεώρηση της νομοθεσίας των διαδικασιών και των πρακτικών που ακολουθεί το δικαστικό σύστημα, καθώς και την υλοποίηση του νέου, κωδικού, του νέου ποινικού κώδικα. Ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να φωτίσουμε τομείς αυτούς όπου ο σεβασμός του κράτους δικαίου μπορεί να ενισχυθεί μαζί με, την, ε, ε, τον πλήρη σεβασμό του συντάγματος του 2008 και τους υπόλοιπους σχετικούς νόμους. Βάσει αυτών των αρχών, οι αρχές των Μαλδιμών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν μια σαφή βάση για να συνεργαστούν περαιτέρω και να προστατεύσουν ε, σε αυξημένο βαθμό το κάτω δικαίου στις Μαλδίβες. Αυτές οι ανησυχίες είναι... συνεχίζονται καθώς υπάρχουν ακόμη εξτρεμιστές που δρούν για να φέρουν τους πολίτες των Μαλδιβών κοντά στις πεπιθήσεις και τις αντιλήψεις των τσιχαντιστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βοηθήσει τις αρχές της χώρας αυτής να αντιμετωπίσει τα πραγματικά αίτια της ριζοσπαστικοποίησης, όμως πραγματική πρόοδος θα εξαρτηθεί καταρχάς από την κυβέρνηση και την έγκαιρη και αποτελεσματική δράση τους για να βεβαιωθούν το πολιτικό σύστημα στις Μαλδίβες είναι όσο το δυνατόν υγιέστερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε, για τη δήλωσή σας αυτή. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το ΕΛΚ. Ο κύριος Στήρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όταν Μιλάμε για τις Μαλδίβες. Η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό των περισσότερων Ευρωπαίων είναι πως μιλάμε για τον παράδεισο επί της γης. Οι ντόπιοι όμως δεν ζουν σε παράδεισο. Είναι πολύ διαφορετικές οι, βιωτικές, ε, οι συνθήκες διαβίωσης ε, και όλο ένα χειροτερεύουν. Για τον Μοχάμετ Νασίτ, πρώην πρόεδρο των Μαλδιβών, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι έχει συλληφθεί και και σε 13 χρόνια ε, κάθερξη, κάτι το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά για το πώς λειτουργεί η δημοκρατία στις Μαλδίβες. Χωρίς να κρίνουμε το κατά πόσο είναι ένοχος ή αθώος, θα έπρεπε να επιμείνουμε στο δικαίωμα που έχει για μια δίκαιη δίκη η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε κομβικό ρόλο το 1998 στον εκδημοκρατισμό των Μαλδιβών όταν ζήτησε να γίνουν δημοκρατικές ε, εκλογές με τον τρόπο αυτό φέρνοντας σε τέλος ε, σε μια δικτατορία 30 ετών. Το 2012 ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος, ο κύριος Νασίτ, παραιτήθηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες. Οι αρχές σήμερα είναι αυταρχικές και δεν συνέχισαν στην πορεία του εκδημοκρατισμού, μοιάζουν να επηρεάζονται από ισλαμιστικές τάσεις και νομίζω ότι αυτός και ένας από τους λόγους που θα ζητήσουμε περισσότερο εκδημοκρατισμό της χώρας αυτής. Θα ήθελα να ζητήσω από την ύπατη εκπρόσωπη Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο μετά στον κύριο Χάουτ για ένα λεπτό. Ενάμιση λεπτό μάλλον. Έχετε το λόγο. Είμαι πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας με την Νότια Ασία και λυπάμαι πάρα πολύ που χρειάστηκε να φέρουμε αυτό το ψήφισμα για τη χώρα αυτή που είναι πανέμορφια νησιά που αντιμετωπίζουν τη μάχη για την κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε όμως να μένουμε σιωπηλοί όταν υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και κάνουμε ό,τι θα κάναμε για οποιονδήποτε κατηγορούμενο που μας δηλώνει πως δεν έλαβε ιατρική φροντίδα, πως δεν έλαβε δικηγορική βοήθεια ή συνήγορο ε, και που δεν ε, αντιμετώπισε μια δική δίκη. Έχει ε, το δικαίωμα οποιοδήποτε να είναι υποψήφιος σε εκλογές παρόλο που στη συγκεκριμένη περίπτωση κατηγορήθηκε για τρομοκρατία με σκοπό μάλλον να αποκλειστεί από τις εκλογές. Το ότι θα στείλουμε παρατηρητές εκλογές νομίζω ότι υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες πως περιορίζονται ε, και, και τα μίντια στη χώρα, αλλά αυξάνονται όλο ένα και οι ένοπλες ομάδες που έχουν πάρει ε, το νόμο στα χέρια τους. Όταν δούμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση και ως μέλος του ΟΕΕ δεν μπορώ να σταθώ σιωπηλός. Ειδικά δε γιατί εγώ ανήκω και στην κοινοπολιτεία. Είναι ο υπουργό Τουρισμού ο ίδιο ο οποίος ανοιχτά δέχτηκε πως κατηγορείται για διαφθορά, βία και τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου. Και στο ψήφισμα αυτό ζητάμε οι συμβολές προς τους τουρίστες από την Ευρώπη να χρησιμοποιηθούν για να ασκήσουμε πίεση. Είναι μια κουκίδα σε ένα τεράστιο ωκεανό. Παρόλα αυτά εξαφανίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορούμε να σταθούμε αδιάφορα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Τάνο. Ένα ε, λεπτό. Η χώρα είναι γνωστή για τον τουρισμό και όχι για ακραία φαινόμενα. Αλλά δυστυχώ οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία επιδεινώνονται στι Μαλδίβε. Αυξάνεται ο σολαφισμό και πολιτικέ εντάσει. Ειρηνικέ διαδηλώσει ε, είναι αντικείμενα διώξεων και το δικαστικό σύστημα χειραγωγείται για να φυλακίζονται αντιπολιτευόμενοι πολιτικού. Η καταδίκη του Μοχάμεν Νασίρ, του πρώην Προέλτου, του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου πρόεδρου των Μαλδιβών, που έκανε τόσο πολλά στο παρελθόν για να αντιμετωπιστεί η άνοδο των υδάτων λόγω τη κλιματική αλλαγή, είναι ένα μόνο παράδειγμα επιλεκτική δικαιοσύνη και διαφθορά σε ένα πολιτικοποιημένο δικαστικό σώμα. Υπόθηκε ότι στη δίκη του δεν τηρήθηκαν ε, οι προδιαγραφές για τη δίκαιη δίκη. Η ομάδα μου καλεί την κυβέρνηση των ε, Μαλτιβών να απελευθερωθεί άνεφορον τώρα ο, πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου. Και τώρα λέγεται ότι θα εισαχθούν και ε, θανατικές πηγές για ανήλικες μέσω της Αρία. Αυτό αυξάνει και την ριζοσπαστικοποίηση σε αυτή τη μικρή χώρα. Το ψήφισμα λοιπόν μας καλεί να αποστείλουμε μήνυμα στους ε, τουρίστες από τις χώρες μας. Μήνυμα προειδοποίησης και επειδή είναι χώρα της κοινοπολιτείας ελπίζω οι Μαλδίβες να επανέλθουν από το χείλο της Αβίσου. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι η κυρία και Δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Το περασμένο μήνα ο κύριος Νασίν, το πρώτος νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος των Μαλδιβών, ε, στάλει και φυλακή, ε, στη φυλακή. Ε, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθεξης. Ε, είναι απαράδεκτα τα γεγονότα αυτά. Καλούμε τις αρχές της χώρας να βεβαιωθούν ότι οι δικαστικές διαδικασίες θα γίνουν βάσει ανεξάρτητων και διεθνών προτύπων, ότι θα έχει συνήγορο πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη εφόσον τη χρειάζεται ο κύριος Νασίν και στους ε, συμβούλους και δικηγόρους με τους οποίους θα πρέπει να μπορεί να συζητήσει. Οι Μαλδίβες είναι ακόμα μια περίπτωση παραβίασης ανθρωπινών δικαιωμάτων με την εξαφάνιση του δημοσιογράφου Αχμέντ ε, ε, Μουνιαμάν, ο οποίος βλέπουμε μαζί με τις διαδηλώσεις που, που, που παρατηρούνται στη χώρα να εντείνει τις ανησυχίες και η αύξηση της προσχώρησης των πολιτών της χώρας αυτής στο τζιχάντ μας ανησυχεί επειδή σε πολλά από τα νησιά αυτά ε, παραθερίζουν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και τουρίστες, θα πρέπει να πιστήσουμε την προσοχή της, Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, σταθερότητα των νήσων αυτών και να φροντίσουμε να υπάρξει ανεξάρτητη εκδίκηση της υπόθεσης του πρώην Προέδρου. Ε, ευχαριστούμε κύριο Σκούσο Περμουή. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε ένα πρόεδρο στη φυλακή, έχουμε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι και αυτοί κρατούμενοι. Όλα αυτά αξίζουν την καταδίκη μας. Και φυσικά το καταδικάσουμε, αλλά πρέπει να τονίσουμε επίσης και ότι υπάρχουν και γεωπολιτικά συμφέροντα τα οποία παίζονται. Τα δύο μετά και δύο σταθμά δεν είναι καυλά για κανένα. Εμείς έχουμε πρώτα προκαλέσει πολέμους εναντίον του Ιράκ, εναντίον της Λιβύης, έχουμε προκαλέσει την αποσταθεροποίηση και της Συρίας. Πολλές φορές τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια φενάκι ώστε η Ευρώπη να εμπλακεί σε διαμάχες που ωφελούν σε εμπορικό επίπεδο την, ε, την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση υποστηρίζει το σχέδιο της Κίνας για τον δρόμο του μεταξιού, αντίθετα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν μιλάμε για πραξικοπήματα και ανθρώπινα δικαιώματα απερίφραστα και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά θα πρέπει να θυμηθούμε τι έκανε η Ευρώπη στην, στη το 2009. Ας μην λοιπόν χρησιμοποιούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πρόσχημα. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Η κυρία Λάμπερτ για ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ μιλώ εξ ονόματο τη ομάδα μου, αλλά είμαι και πρόεδρο τη αντιπροσωπεία με την Νότια Ασία που περιλαμβάνει και τι Μαλβίδε. Μια χώρα που επισκεφθήκαμε μετά από το τσουνάμι και στην εποχή που συζητεί το ακόμα το νέο σύνταγμα, κάτι το οποίο υποστηρίξαμε στις Μαλδίβες. Η νεαρή δημοκρατία των Μαλδιβών έχει προχωρήσει σε κάποιο βαθμό στον δρόμο της δημοκρατίας, αλλά υπήρξαν και πολλές εντάσεις σε ό,τι αφορά την εγκαθίδρυση νέων θεσμών εκεί. Ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλος του που διαδραμάτισε ο προηγούμενος πρόεδρος Ασίτ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκφράσει και την ανησυχία του όταν ως πρόεδρος ζήτησε να συλληφθεί ένας δικαστικός, κάτι το οποίο είχε σημαντικές ε, επιπτώσεις. Τα πρόσφατα γεγονότα είναι πραγματικά ανησυχητικά βλέπουμε να χρησιμοποιείται η αντιτρομοκρατική νόμοι χωρίς να δίνεται το δικαίωμα στους κρατούμενους να χρησιμοποιήσουν το συνταγματικό δικαίωμα της ε, υπεράσπισης. Υπάρχει αλλαγή στο νόμο για τα τη συμμετοχή σε δημόσια αξιώματα και οι διαδικασίες δικαστικές δεν επιτρέπουν την προετοιμασία μιας έφεσης. Με μεγάλη δυσκολία μπορώ να φανταστώ ότι όλα αυτά είναι απλώς μια απλή σύμπτωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εξασφαλιστούν οι συνταγματικές εγγυήσεις στις Μαλδίβες για όλους τους πολίτες είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το μικρό νησί, το οποίο επιπροσθέτω απειλεί και από την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Οι μεμονωμένοι ομιλητέ, ο κύριο Πρέντα πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρα. Ο Μοχαμέτ ε, Ρασίδ, Νασίδ, ο πρώην πρόεδρο των ε, Μαλδιβών, συνελήφθη πριν από 1,5 χρόνο για 8η φορά σε 25 χρόνια. Υπήρξε σύμβολο της δημοκρατίας στις Μαλδίβες, στη χώρα του και μετά από χρόνια μη βίαιης αντιπολίτευσης πέρασε φυλακή, εξορία και το 2008 έγινε ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος του νησιού, θέτοντας τέρμα σε 30 χρόνια του Μαμούν Αμπτούλ Γκαϊού ανάληψη της εξουσίας μετά από ελεύθερες εκλογές ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη δημοκρατικοποίηση της χώρας αυτής. Δυστυχώς αυτό δεν ήταν επαρκές. Η πολιτική κατάσταση στις Μαλδίβες είναι παραπάνω από ανησυχητική γιατί οι κρατικοί θεσμοί είναι πολιτικοποιημένοι και αυτό περιλαμβάνει και το δικαστικό σύστημα. Οι κατηγορίες για τρομοκρατία κατά του Νασίρ που επισύρουν 13 χρόνια φυλακή, φυλακίσεις δείχνουν ότι η φυλακή, ότι η δικαιοσύνη, συγγνώμη, την χάνει εκμετάλλευση από τις πολιτικές αρχές. Η οικογένεια Γκαγιούμ έχει πάλι την εξουσία γιατί ο τωρινός πρόεδρος είναι γαμπρός της προηγούμενης αυτής οικογένειας και η κόρη της οικογένειας είναι ο υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Είμαστε πολύ μακριά από το δημοκρατικό καθεστώς το οποίο είχαν επιλέξει οι πολίτες των Μαλδιβών το 2008 και ψήφισαν γι' αυτό. Είναι απαραίτητο λοιπόν να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στις Μαλβίδες. Ο κύριος Μόσκα. Κυρία Μόσκα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε πολλά μέρη του κόσμου βλέπουμε ε, τέτοιες καταστάσεις και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να είμαστε αναίσθητοι και αδρανείς σε σχέση με αυτές τις καταστάσεις. Η πολιτική κατάσταση απειλείται, απειλείται το κράτος δικαίου. Γι' αυτό η προσοχή μας στρέφεται πριν απ' όλα στην νοικοδόμηση ενός ειρηνικού κλίματος και μιας νυφάλιας πολιτικής συζήτησης με στήριξη έτσι ώστε η αστυνομία να δεσμευτεί και να προστατεύσει την ε, ελευθερία του διαδηλώνων με πάσα ασφάλεια ε, μέχρι σε ότου να αποπολιτικοποιηθούν οι δικαστικές αρχές. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σρι Λάγκα και τις Μαλδίβες θα παρακολουθεί την κατάσταση παρέχοντας στην ύπατη εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη όλες τις πληροφορίες και τα μέσα για να δράσει ε, ε, ε, με όλα τα διμερή και διεθνή μέσα για να αποκατασταθεί το δημοκρατικό σύστημα στις Μαλδίβες και να εξασφαλιστεί ο συμβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρουντζουλίτσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι οι Μαλδίβες δεν είναι πια μόνο ένας ε, τουριστικός παράδεισος. Έχουν μετατραπεί σε ένα μέρος όπου ε, αυξάνεται ο κίνδυνος λόγω φονταμενταλιστών μέσω ενός πολιτικοποιημένου δικαστικού συστήματος και της διάβρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Στη μένη δίκη του πρώην Προέδρου Μοχάμετ Νασίρ δείχνει πώς ε, πόσα προβλήματα υπάρχουν εκεί για τη δημοκρατία. Αυτή η υποτιθέμενη δίκη δεν σέβεται τους βασικούς κανόνες για δίκαιη δίκη και είναι αντίθετη με το σύνταγμα του κράτους. Ανέκαθεν εμείς στηρίζαμε την ε, σταθεροποίηση της δημοκρατίας, προωθούσαμε την καλή διακυβέρνηση, ενισχύαμε τα, τους θεσμούς και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις Μαλδίβες να αντιμετωπίσει όλες αυτές οι προκλήσεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε ρόλο στη δημοκρατική μετάβαση της χώρας, επισήμως καλώντας για τέλος της βίας κατά των ειρηνικών διαδηλωτών και εξασφαλίζοντας ε, πλήρως ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων του κύριου Νασίρ και την προσήλωση των Μαλδιβών στα διεθνή πρότυπα. Σας ευχαριστώ. Φτάσαμε τώρα στο τέλος αυτής της ε, συζήτησης με τους μεμονωμένους ε, ομιλητές και θα προχωρήσουμε με τη διαδικασία Catch the Eye, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δώσω το λόγο σε όλους όσους το ζήτησαν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, ήμουν επικεφαλής της ε, αποστολής για να παρατηρήσουμε τις εκλογές στις Μαλδίβες. Ήταν ειρηνικά τα πράγματα ε, και διεξήχθηκαν οι εκλογές με επαγγελματικό τρόπο. Ε, κι όμως δύο μέλη της Επιτροπής Εκλογές απομακρύνθηκαν από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ήταν νομίζω παραβίαση της αρχής του διαχωρισμού των εξουσιών και της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Εκλογών. Ε, μετά από ένα χρόνο έχουμε αμφισημίες με το θέμα του Πρόεδρου Νασίντ. Κάθε δημοκρατική χώρα πρέπει να σέβεται τις νομικές διαδικασίες, το σεβασμό του κράτους δικαίου και την ανεξαρτησία του, της δικαστικής εξουσίας. Δεν είναι η περίπτωση με το θέμα Νασίντ. Θα μπορούσαμε να στείλουμε παρατηρητές στην δίκη του Νασίντ, εάν αποφασίσει να κάνει έφεση. Ο κύριος Μαριάς ζήτησε το λόγο. 13 Παρτίου του Μουχάμετ Νασίτ, του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου των Μαλδιβών, ενός, ενός ανθρώπου που έχει ταχθεί υπέρ της μη άσκησης βίας και η καταδίκη του σε 13 χρόνια φυλάκιση αποτελεί αποκορύφωση του περιορισμού της δημοκρατίας στις Μαλδίβες ακολούθησαν και άλλες αποφάσεις του κοινοβουλίου της χώρας αυτής που περιορίζουν τα δημοκρατικά δικαιώματα τη δραστηριότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δημοσιογράφων. η κατάσταση λοιπόν στη χώρα αυτή είναι κρίσιμη και τα πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν την ανάγκη για βαθιές δημοκρατικές αλλαγές. απαιτείται λοιπόν η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος η αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και ο σεβασμός της ελευθερίας έκφρασης και συνάθρησης η πλουραλιστική δημοκρατία στις μαλδίβες πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει και να κλείσει ο δρόμος στους τζιχαντιστές. γι' αυτό η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της ελευθεροτυπίας και στη λειτουργία του κράτους δικαίου στις μαλδίβες. Η Ευρώπη έχει κάνει πολλά για τις Μαλβίδες με πολλούς τρόπους και οικονομικά και πολιτιστικά και πολιτικά. Ξέρουμε ότι το νέο σύνταγμα του 2008 άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία των Μαλδιβών. Ξέρουμε ότι έχει πράξει και η Ευρώπη για αυτό το κράτος επίσης. Αλλά η δημοκρατία ήταν βραχίδια. Δεν ε, λαμβάνω το λόγο για να αναφερθώ στο αν η τωρινή ηγεσία της, ε, των ε, Μαλδιβών είναι υπέρ του Ισλάμ ή υπέρ της Κίνας. Αλλά ξέρουμε ότι ο προηγούμενος, ο πρώην πρόεδρος, έχει το δικαίωμα σε μια δίκαια δίκη, έχει κάθε δικαίωμα σε ιατρική φροντίδα και περίθαλψη <clears throat> και θα πρέπει να πούμε ανοιχτά ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να προστατευτεί από τη δικαιοσύνη. Κύριος Γκαστάλτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει μια ανησυχητική πραγματικότητα στι Μαλδίβε που οι γυαλιστερέ σελίδε των τουριστικών καταλόγων δεν διηγούνται. Σήμερα ακριβώ γίνονται όλα αυτά με το καταδίκη του πρώην Πρόεδρου Μοχαμέτ Νασίρ σε 13 χρόνια κάθριξη. Πολλοί διεθνεί παρατηρητέ λένε ότι πρόκειται για πολιτική φάρσα, όπω είπε και η, η Διεθνή Αμνηστία. Εχθέ διαδήλωσαν φτάνοντας στην πρωτεύουσα με ε, βάρκες. Δυστυχώς όμως συνελήφθησαν και εκφοβίστηκαν δημοσιογράφοι ώστε να μην ε, συνεχίσουν. Η χώρα ταξιδεύει σε τελείως διαφορετικό δρόμο. Ε, <laughs> ισχύει ακόμα η θανατική ποινή. Ακόμα και παιδιά 13 χρονών ε, μπορεί να δικαστούν. Ε, στις ε, η πρώτη απειλή είναι η κλιματική αλλαγή και, και αυτό έχει ξεχαστεί. Πιστεύω πως πρέπει να δεσμευτούμε εντόνως ώστε η νέα αυτή εκτελεστική κυβέρνηση να μην ε, θεωρεί πως το κράτος δικαίου είναι προαιρετικό αυτός ο παράδεισος των διακοπών να μην μετατραπεί σε κόλαση της δημοκρατίας. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω τους προλαλήσαντες που αναφέρθηκαν στην κατάσταση στις Μαλδίβες. Οι δικαστικές διαδικασίες έδειξαν ότι ο πρώην ε, πρόεδρος ε, καταδικάστηκε. Δεν είχε δίκαιη δίκη και το θέμα της ρίζοσπαστικοποίησης στις Μαλδίβες είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να μας ανησυχεί. Θα πρέπει να λέμε σε όλους τους τουρίστες ε, οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν αυτόν τον παράδεισο των νησιών ότι η τουριστική ε, δραστηριότητα προωθείται ε, στις, ε, στα φυλάδια, αλλά η κατάσταση εκεί δεν είναι ίδια. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κυρία Μογκερίνη και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μην ακολουθηθεί το, παράδειγμα της ISIS. Έχουμε το τέλος του, της διαδικασίας Catch the Eye και δίνω τον λόγο στον κύριο Μίμητσα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Ευχαριστώ για τη συζήτηση που τόσο σαφώς εξέφρασε την υποστήριξη στη δημοκρατική διαδικασία και στο σεβασμό του κράτους δικαίου στις Μαλδίβες. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στις Μαλδίβες. Ε, νομίζω ότι η εξωτερική δράση και η αντιπροσωπεία που βρίσκεται στο Σρι Λάνκα και καλύπτει τις Μαλδίβες θα παραμείνει σε στενή σχέση με την κοινωνία των πολιτών, με τους πολιτικούς παράγοντες. Περιμένουμε η κυβέρνηση των Μαλδιβών να δεχθεί τις προτάσεις, τις πολιτικές και νομικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες θα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Μαλδίβες την ευκαιρία να αρχίσουν ένα διάλογο για την κατάσταση της δικαστικής εξουσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την Ισλαμική ριζοστικοποίηση που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου θα θέλαμε να βοηθήσουμε τις Μαλδίβες και τον πληθυσμό να έχουν μια δημοκρατία που να τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη δέσμευσή σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Λεκή Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στον, ε, στην Κομισιόν. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουν υποβληθεί επτά ψηφίσματα τα οποία θα ψηφιστούν αργότερα. Φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης και θα ψηφίσουμε αύριο για το θέμα αυτό.